So, Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές συνάδελφοι, μεγάλη χαρά και τιμή για μένα σήμερα ως πρώην πρόεδρος της Επιτροπής, ως τέος πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού, σας καλωσορίζω. Εδώ βλέπω πολλά γνώριμα πρόσωπα, αλλά και μία σειρά νέων προσώπων. Σας καλωσορίζω όλους θερμά και ελπίζω και οι εργασίες σας στην Επιτροπή Πολιτισμού για την επόμενη πενταετία να στεφθούν με επιτυχία και να χαρακτηριστούν από μια επικοδομητική συνεργασία όπως άλλωστε και τα προηγούμενα πέντε, για να μην πω τα τελευταία δέκα χρόνια που είμαι εγώ εδώ σε αυτή την Επιτροπή. Κυρίσω λοιπόν την έναρξη συνεδρίασης. Πρώτα απ' όλα. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους τους βουλευτές ότι έχουμε μετάδοση μέσω του διαδικτύου, Webstream της συνεδρίασης. Σήμερα ε, θέμα μας είναι η συγκρότηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Εκπαίδευσης, ε, εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρων, όπως ορίζει το άρθρο 213 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου. Έχουμε την εξής σειρά. Πρώτα εκλέγεται ή ή ο Πρόεδρος και στη συνέχεια ένας-ένας οι αντιπρόεδροι της Επιτροπής. Διερμηνία έχετε σήμερα σε όλες τις επίσημες γλώσσες, πλην της δανικής λέει η πρόεδρος. Εμείς βλέπουμε τους δανούς συναδέλφους εδώ, δεν υπάρχουν όμως, και της κελτικής. Και γίνεται η εκλογή λοιπόν τύση του Προέδρου και στη συνέχεια των αντιπροέδρων με τους αντικαταστάτες Σόφκο για τον κύριο Άντιμοφ, Μπέρν Χουμπεα που αντικαθιστά τον κύριο Πόλακ, τον κύριο Κόχουτ που αντικαθιστά τον κύριο Χάιντε, τον κύριο Κόλαγια που αντικαθέτω τον κύριο Νίσας και την κυρία Ντέμπο Σκόφιλτ που αντικαθέτω την κυρία Ζαμπού την κυρία Μπαλτάσαρ που αντικαθέτω τον κύριο Τζαναντώνιο και τον κύριο Μουμπάρικ που αντικαθέτω τον κύριο Σλάμπακοφ. Έχετε κάποιον άλλον ε, που πρέπει ως αναπληρωτές να αντικαταστήσετε. Κύριο Πόλακ, ναι. Είναι εδώ από ό,τι βλέπω μάλιστα. Καλώς. Άρα, διαγράφουμε το όνομα του αναπληρωτή. Έχετε κάποιον άλλον που πρέπει να αντικατασταθεί από τον αναπληρωτή του, τακτικό μέλος που αντικαθίσταται, όχι. Καλώς. Και θα ήθελα να ενημερώσω τις ομάδες που σε περίπτωση ε, τροποποίησης ε, πρέπει να ενημερώσουν την ε, πρόεδρο, την προεδρεύουσα κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας αν υπάρχει κάποια αλλαγή σε σχέση με τη σύνθεση. Πρέπει να κοινοποιηθεί στην γραμματεία. Η απαρτία είναι δεδομένη, χρειάζονται τουλάχιστον 8 συνάδελφοι. Προφανώς λοιπόν μπορούμε να λάβουμε τη σχετική απόφαση με τις ψηφοφορίες και παρακαλώ τώρα να μου πείτε ποιοι είναι οι υποψήφοι για την θέση του ή της Προέδρου, κυρία Σόντροβα πρώτη. Πρόεδρε, καλημέρα σας. Έχω την τιμή και χαρά να προτείνω εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος την κυρία Φων τη συνάδελφο ως πρόεδρο της Επιτροπής Κούλτ. Κυρία Κάμερεβερτ, ευχαριστώ. Η Ζαμπίνα Φερχάιεν είναι τακτικό μέλος της Επιτροπής, υποψήφια εκ μέρους της ομάδας της. Την ερωτώ αν έχει καταθέσει τη σχετική δήλωση για τα οικονομικά συμφέροντα και την ε, δεοντολογία. Όλα αυτά έχουν τακτοποιηθεί, πολύ ωραία εξαίρετα. Και ερωτώ αν υπάρχουν και άλλοι υποψήφοι για τη θέση του Προέδρου. Προφανώς όχι και ερωτώ εάν η Ζαμπίνε δέχεται βέβαια καταρχάς την ε, υποψηφιότητα αυτή. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν μία υποψήφια για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Πολιτισμού και ερωτώ εάν δέχεστε διαβοής να ανακηρύξουμε την Ζαμπίνε Φερχάιεν ως Πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτισμού. Ζαμπίνε, Φαντάζομαι ότι δέχεσαι την εκλογή σου και σε παρακαλώ να έρθεις στο Προεδρείο να καταλάβεις τη θέση σου. Du bringst die Blumen schon selber mit. Δυστυχώ η ομιλία τη κυρία Φερχάιν δεν ακούγεται, διότι δεν υπάρχει μικρόφωνο αναμένο στην αίθουσα. I also would like to say thank you. Και στα αγγλικά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους και όλες για την εμπιστοσύνη που μου δείχνετε στην αρχή αυτή της θητείας μας και ελπίζω πως όπως και στο παρελθόν θα έχουμε πολύ καλή και επικοδομητική αλλά και ειρηνική συνεργασία στην Επιτροπή μας. Είχαμε πάντα καλή συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια. Μέλος της Επιτροπής είμαι εδώ και πολλά χρόνια. Ως τακτικό μέλος, συντονίστρια πάντα είχα με τιμή να επιτελέσω το έργο μου. Τώρα και ως Πρόεδρος συνεχίζω να προσφέρω τις υπηρεσίες μου σε αυτή την συνεδρία, στην Επιτροπή, στην οποία πάντα συνεργαζόμαστε με πολύ φιλικό τρόπο. Και τώρα, Ψηφίζουμε τον πρώτο ή την πρώτη αντιπρόεδρο. Ενημερώθηκα πως ε, έχουν κατατεθεί τα εξής ως πρόταση για του αντικαταστάτε, αναπληρωτέ τακτικών μελών. Αυτό ανακοινώθηκε νωρίτερα από την κυρία Καμερέβερτ. Ερωτώ λοιπόν αν υπάρχει κάποια αλλαγή εντωμεταξύ στι ε, αναπληρώσει τακτικών μελών. Όχι. θα ήθελα να ενημερώσω ότι πριν από κάθε επιμέρους ψηφοφορία θα πρέπει πάντα να σας ερωτώ εάν έχει αλλάξει κάτι στη σύνθεση των μελών, δηλαδή στην εκπροσώπηση. Εφόσον λοιπόν δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, δεν αλλάζει και η απαρτία μας που ήταν ε, με ελάχιστα 8 μέλη και παρακαλώ να μου πείτε ποιος ενδιαφέρεται να δηλώσει ε, πώς προτείνει για υποψήφιο αντιπρόεδρο. Καλημέρα σας για τη θέση του πρώτου αντιπροέδρου. Θα ήθελα να προτείνω τον κύριο Γόμεο Φραντς εκ μέρου των Πρασίνων Ελεύθερης Συμμαχίες. Ελεύθερης Πράσινης Συμμαχίας. Μάλιστα, ο κύριος Γόμεο Φραντς προτείνεται με βάση το σύστημα DONT. Πρόκειται άλλωστε για θέση που αντιστοιχεί στους Πρασίνους. Τακτικό μέλος της Επιτροπής ε, από τους συναδέλφους του προτείνεται. Έχει καταθέσει σχετικές δηλώσεις οικονομικών ε, συμφερόντων και δεοντολογίας. Έτσι δεν είναι, μάλιστα. Και σας ερωτώ, κύριε υποψήφιε, εάν το δέχεστε. Βεβαίως, δέχομαι την υποψηφιότητα. Καλώς, υπάρχει άλλος υποψήφιος. Όχι από ό,τι βλέπω. Και δεδομένου ότι έχουμε μόνο έναν υποψήφιο, παρακαλώ να επικροτήσουμε τον κύριο Ρώμεο Φραντς στη θέση αυτή διαβοής Σας εύχομαι και εγώ κάθε επιτυχία, κύριε Φραντς, και αγαστή συνεργασία στην Επιτροπή μας. Περάστε παρακαλώ στο Προεδρείο να καθίσετε στη θέση σας. So, dann kommen wir nun zum, zur Wahl des zweiten stellvertretenden Vorsitzenden. Auch hier muss ich noch mal wieder Περνώ στην εκλογή τώρα δεύτερου αντιπροέδρου. Διαπιστώρω και πάλι ότι δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στη σύνθεση των μελών που θα ψηφίσουν εδώ. Ε, οι ομάδες παρακαλώ να έχουν υπόψη ότι πριν από την ε, ψηφοφορία πρέπει πάντα να ενημερώνουν αν τυχόν και αλλάξει κάτι στη σύνθεση. Η απαρτία είναι εξασφαλισμένη και πάλι και πάντα. Και παρακαλώ τώρα να ακούσουμε υποψηφιότητες για τη θέση του δεύτερου αντιπροέδρου. Το σύστημα DONT προβλέπει πως πρόκειται για ε, θέση που θα αντιστοιχούσε στην ομάδα ECR. Εκ μέρους της ομάδας ECR θα ήθελα για τη θέση του δεύτερου αντιπροέδρου να προτείνω τον Τάτσι Πάρτι που είναι πρώην υπουργό Πολιτισμού της Λετωνίας και διευθύντρια συγγνώμη, του Κέντρου Πολιτισμού στη συνέχεια. Έχει διατελέσει και υφυπουργό ε, και γραμματέας στο Υπουργείο Πολιτισμού, γενική γραμματέα στην ε, Λετωνική ε, Γενική Γραμματεία της UNESCO και έχει, κάνει, έχει διατελέσει και αντεπιστέλων μέλος μεταξύ Λετωνίας και UNESCO. Σας ευχαριστώ, νέο μέλος του Κοινοβουλίου. Χαιρόμαστε που υποβάλλετε την υποψηφιότητά σας κυρία Ντάτσι Μιλμπάτη, κάπω έτσι, δεν ξέρω αν το πρόφερα σωστά, αν όχι διορθώστε με. Τακτικό μέλος ε, είστε της Επιτροπής, ε, σας πρότεινε η ομάδα σας στο ECR, δήλωση χρηματοοικονομικών συμφερόντων ε, και σε ό,τι αφορά τον κώδικα διοντολογίας έχει κατατεθεί, συμπληρώθηκε, μπορείτε να το επιβεβαιώσετε αυτό. Ναι, βεβαίως. Θέλω να ρωτήσω την υποψήφια να μας πει αν συμφωνεί με την υποψηφιότητα. Ναι, βεβαίως, με μεγάλη χαρά. Πρόεδρος, και εδώ έχουμε μόνο μία υποψηφιότητα. Προτείνω λοιπόν να, εγκρίνουμε την δεύτερη αντιπρόεδρο διαβοής. Ja, dann darf ich Συγχαρητήρια για την εκλογή σας ε, και προσβλέπω σε μια πολύ καλή επικοδομητική συνεργασία και με εσάς. Σας παρακαλώ, ελάτε να καθίσετε στο Προεδρείο. Wir hätten jetzt einen dritten und vierten Stellvertreter. Πρέπει να εκλέξουμε τρίτο και τέταρτο αντιπρόεδρο αλλά υπήρξαν κάποιες συζητήσεις ε, σε ό,τι αφορά ε, την αποδοχή των υποψηφιωτήτων με βάση το σύστημα ΔΕΟΝΤΑ. Θα έλεγα λοιπόν να διακόψουμε τώρα εδώ τη διαδικασία της ε, ψηφοφορίας και να συνεχίσουμε στην επόμενη συνεδρίαση ώστε να έχουμε τη δυνατότητα στο μεταξύ να συζητήσουμε και να καταλήξουμε. για να μην ξεκινήσουμε άσχημα τις εργασίες της ε, Επιτροπής μας, ώστε να έχουμε καταλήξει λοιπόν σε λογικούς ορισμούς. Σήμερα μόλις το πρωί προέκυψε αυτό το πρόβλημα σε ό,τι αφορά τον ορισμό υποψηφιωτήτων. Υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις δηλαδή από ορισμένους συναδέλφους. Γι' αυτό θα σας παρακαλέσω, ή μάλλον δεν σας παρακαλέσω, θα ε, διακόψω σε αυτό το σημείο την διαδικασία και θα την συνεχίσουμε στην επόμενη συνεδρίαση. Η Πέτρα, καταρχήν δεν έχω κάποια αντίρρηση, γιατί και εγώ θεωρώ ότι καλό θα ήταν να κάνω μια πολύ καλή εκκίνηση, μια ομαλή εκκίνηση. Ε, δεν ξέρω κατά πόσον ε, αυτό προβλέπεται από τον εσωτερικό κανονισμό και τι γίνεται συνολικά με την συγκρότηση σώμα της Επιτροπής. Δηλαδή δεν συγκροτείται σε σώμα η Επιτροπή μας και πρέπει να περιμένουμε γιατί αυτό δεν θα ήταν ίσως καλό να συμβεί. Also es ist so, dass die äh, äh Geschäftsordnung des είναι επιτρεπτό. Ήδη έχει συγκροτηθεί η Επιτροπή μας σε σώμα, εφόσον εκλέξαμε πρόεδρο και δύο πρόεδρους. Υπάρχει δυνατότητα της αναβολής, ε, της συνέχισης της διαδικασίας. Αυτό ε, πρότεινα, όπως είπα, για να επιτρέψω να έχουμε μια ομαλή εκείνη των εργασιών μας. Και την μέθε επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες έχουμε εδώ συνεδρίες και εκεί μπορούμε να συνεχίσουμε ε, τη διαδικασία. Αλλά ε, πρώτα να ψηφίσουμε. Υπάρχει κάποιος που είναι αντίθετος με την πρόταση αυτή. Αποχές υπάρχουν, αν όχι... Η εκλογική διαδικασία αναβάλλεται για την προσεχή συνεδρία της Επιτροπής μας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στις 23 Ιουλίου στις 9 το πρωί. Από τις 9 έως τις 12 και μισή και από τις 3 έως 6.30 το απόγευμα ή όχι. Το απόγευμα δεν ξέρω. Λοιπόν, α, έχουμε και κάποια άλλα σημεία. Να σας ενημερώσω ότι την επόμενη Δευτέρα στις 15 Ιουλίου έχουμε μια πρώτη συνάντηση των συντονιστών στο Στρασβούργο από τις 7 9 το βράδυ. Επίσης υπάρχει ένα πακέτο υποδοχής, ένα welcome pack, το οποίο θα σας δώσει κάποιες πληροφορίες ενημερωτικές και σημαντικές πληροφορίες σε σχέση με τις προηγούμενες εργασίες της Επιτροπής μας. Αυτά ε, τα έγγραφα, αυτά τα φυλάδια θα τα βρείτε στη, στη ρίδα σας, ε, στον τρίτο όροφο, για να ενημερωθείτε. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τους διερμηνείς και, όπως είπα, προσβλέπω σε μια επικοδομητική μελλοντική συνεργασία και σε μια ομαλή ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας της 23 του μηνός. Ευχαριστώ πολύ.